ενημερώνει για αυτήν την αντικατάσταση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά αυτή την αντικατάσταση. Όχι, λοιπόν, θεωρούμε ότι ο κύριος Σόλτς παίρνει τη θέση του κύριου Γκούσταυσον. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 4, θα ήθελα να σας ε, ανακοινώσω ότι θα τεθεί σε ψηφοφορία το κείμενο το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα Seance on Direct και έχει δημοσιευθεί την Τρίτη σύμφωνα με το άρθρο